Καλησπέρα σας. Όπως σας είχα υποσχεθεί και το πρωί και σας θερμό παρακάλεσα, θα αρχίσουμε αμέσως, α, ακριβώς την ώρα μας, είναι τρεις και κάτι. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Γκίντερ Ότιγκερ, που είναι αρμόδιο για τον προπολογισμό και του ανθρώπινους πόρους για μια ανταλλαγή απόψεων επί του εγγράφου προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, βέβαια, είναι πολύ άσχολος ο Επίτροπο τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να συναντηθεί με πολλούς, να ακούσει διάφορες πληροφορίες. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι οι συντονιστές θα έχουν από δύο λεπτά ο καθένας και από δύο λεπτά επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές γιατί είναι μετρημένος ο χρόνος μας. Γι' αυτό και δεν θα κάνω καμία άλλη εισαγωγή. Θα δώσω αμέσω το λόγο στον επίτροπό μας, τον κύριο Έτιγκερ, για να μας κάνει την παρουσίασή του. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε στην σημαντική επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται στην παρούσα χρονική στιγμή για την χορήγηση συμβουλών, τη διατύπωση προσδοκιών σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου για την επόμενη δεκαετία. Πού βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως και εσείς και εμείς αντιμετωπίζουμε τη μελλοντική γεωργική πολιτική με ανησυχία. Καταρχάς, θέλουμε να υποβάλουμε ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο και πάλι. Γιατί τα επτά έτη σημαίνει νομική δεσεβαιότητα και ασφάλεια για όλες τις εμπλεκόμενες φορείς, ε, για τους ε, αγρότες, τους νεαρούς αγρότες, τους ε, καταναλωτές στην Ευρώπη αλλά θέλουμε να ανακοινώσουμε ότι η μεθεπόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι πενταετές ή πέντε συν πέντε έτη. Γιατί τότε το, το 2024 θα εκλεχθεί κοινοβούλιο, το Μάιο. Το Νοέμβριο του 2024 θα ξεκινήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θετία της και για ένα τμήμα της ε, δικής της θητείας θα μπορέσουν ε, και τα δύο σώματα να αποφασίσουν ε, για την προεπλογισμό τους. Και έτσι λοιπόν στο με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει μεγαλύτερη αντιστοιχία με τη θητεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά δεύτερον, θέλουμε ένα κοινό πλαίσιο για την κοινή πολιτική στο μέλλον. Κατά τρίτον, φυσικά υπάρχουν επιχειρήματα να συνδυαστεί ο δεύτερο πυλώνα με την πολιτική συνοχή. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχουν και σημαντικά επιχειρήματα για τη διατήρηση των δύο πυλώνων στο εσωτερικό της κοινή ε, γεωργική πολιτικής. Προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία στην Επιτροπή σας, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά να μείνουν στην αρμοδιότητα δική σα, λοιπόν. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, λοιπόν, τα θέματα αρμοδιότητα, το πώ θα κατανείμουμε τα μέσα μεταξύ τη πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Τώρα έχουμε και το άλλο αποφασιστικό ζήτημα. Έχουμε δύο δημοσιονομικά κενά στο επόμενο που το πω. Το πρώτο κενό είναι το Brexit. Ένα χάσμα που προκύπτει από έλλειμμα προσόδων, εσόδων. 12 έως 13 δις ευρώ θα μας λείψουν κάθε χρόνο δομικός πώς. Και έχουμε και, και ένα κενό σε ό,τι αφορά τις δαπάνες και τα καθήκοντα. Γιατί σε σύγκριση με τις διαβουλεύσεις ε, του τρέχοντος ε, Πουδουπού 2011-2012-2013, την επόμενη δεκαετία θα υπάρξουν νέα καθήκοντα, τα οποία θα μπορούμε καλύτερα και με πιο ευνοϊκό κόστος να τα κοιτάξουμε σε κάποιες περιπτώσεις και μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα των προσφύγων. Αναπτυξιακή βοήθεια για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, έλεγχο συνόρων και προστασία συνόρων, μετανάστευση, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, έρευνα. Έρευνα άμυνας και βιομηχανία της άμυνας. Θεωρούμε, παρά το γεγονό ότι αυτές οι δαπάνες και τα καθήκοντα αυτά δύσκολα εκτιμώνται, μόνο ένα τμήμα αυτών άλλωστε περιλαμβάνεται στο τρέχον πουδουπού, θεωρούμε ότι μέσω ευελιξίας μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε στο ιστορικό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά τα καθήκοντα αυξάνονται και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται στο προπολογισμό, να υπάρχει επαρκή χρηματοδότηση που να προβλέπεται στο επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, επί της αρχής είμαστε κατά των περικοπών σε ό,τι αφορά την κυνηγεργική πολιτική. Εμείς εργαζόμαστε για δύο-τρεις τύπους που θα πρέπει να διαμορφώνονται στο, στη διαμορφωσή του προπολογισμού. Το κενό του Brexit, το θέμα του 50% μέσω μείωση των τρέχουσών δομών του προπολογισμού και 50% καινούργια χρήματα. Το κενό που προκύπτει από τις νέες δαπάνες και από τα νέα καθήκοντα που θα είναι προς το όφελος των κρατών μελών και των πολιτών είναι 80% από καινούργια χρήματα θα καλυφθεί και μόνο 20% θα καλυφθεί από ανακατατάξεις στην υφιστάμενη δομή του προϋπολογισμού. Και αν τα προσθέσουμε όλα αυτά με πάσα σοβαρότητα, τα υφιστάμενα προγράμματα συνοχή, ΚΑΠ, διευκολύνοντας την Ευρώπη, ορίζοντας 2020, Erasmus Plus και άλλα τέτοια μεγάλα προγράμματα. Και αν τα νέα καθήκοντα τα αποτυπώσουμε με ρεαλιστικό τρόπο στο προϋπολογισμό, θα χρειαστούμε ένα ανώτατο όριο για την πλευρά των εσόδων και για τις δεσμεύσεις 1,1 χ. Και βάζουν το χ από 1,11 έως 1,19 εννοώ. Το Κοινοβούλιο προετοιμάζει στην παρούσα φάση δύο καινούργιε εκθέσει. Η κυρία Τόμα και ο κύριο Όλμπρεχτ, οι συνάδελφοί σα, ε, Ντεπρέ και Λεοντόφσκι, είναι οι αρμόδιοι εισηγητέ και προσβλέπω στη συζήτηση το Μάρτιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα προτείνει κατά πάσα πιθανότητα το 1,3% ως ανατοτόριο. Ως εδώ έχει καλώς. τα τελευταία... Ε, έχω πάει ήδη σε 17 κράτη-μέλη και θα πάω και στα 10. Έχω συνομιλήσει με τους υπουργούς εξωτερικών, οικονομικών, με τους πρωθυπουργού, με τα εθνικά κοινοβούλια στα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ωστόσο ότι 5-6 κράτη-μέλη θα υπάρξουν, τα οποία θα προασπίσουν αμετακίνητα τη γραμμή του τρέχοντος ε, πουδουπού, το οποίο το είχε προασπίσει και ο David Cameron, το 1,0% ως ανώτατο όριο. Αμετακίνητα. Σουηδία, Φινλανδία, Δανία, κάτω χώρες, Αυστρία. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στην Επιτροπή, υπάρχουν βουλευτές από τις χώρες αυτές, οι οποίοι φαντάζομαι θα επιβεβαιώσουν πόσο αμετακίνητη είναι η Στοκόλμη, η Κοπεχάγη, η Χάγη, για, η Βιέννη για το 1,5%. Αυτό απλά το σημειώνω, το λαμβάνουμε υπόψη. Αν υπάρχει αυτό είναι το σημείο φετηρία της συζήτηση έχει καλώς. Αν αυτή είναι όμως η τελική θέση, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Γιατί με το 1,0% χωρίς τα αφιστάμενα μεγάλα προγράμματα, μάλλον χωρίς να βλάψουμε τα μεγάλα μας προγράμματα, τον ορίζοντα, το Εράσμους, την ΚΑΠ λοιπά, δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να εκπληρώσουμε με σοβαρό τρόπο και να χρηματοδοτήσουμε τις παλιέ και τις νέε ε, αρμοδιότητες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε στο 1,1 χ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εσείς ως αρμόδια επιτροπή είσαστε κατά των περικοπών. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν θα εμείνετε στη θέση σας αν ε, τυχόν ε, χρειαστεί να γίνουν περικοπές. Παρ' όλα αυτά, να μου πείτε πού μπορούν να γίνουν και πού δεν μπορούν να γίνουν περικοπές, χωρίς τη δική σας ε, θέση. Χωρίς να απαρνηθείτε τη θέση σας ότι δεν θέλετε τις περικοπές επί της αρχής. Με το έγγραφο περισυλλογής, με την ανακοίνωση για το ανεπίσημο, την ανεπίσημη σύνοδο που θα λάβει η χώρα στις ε, Βρυξέλλες και με συζητά, πώς συζήτηση με τον συνάδελφο Χόγκαν, διαμορφώσαμε κάποιες σκέψεις και τις δημοσιεύσαμε. Τον Απρίλιο, λοιπόν, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ορίσουμε οριστικά τις ε, θέσεις μας σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το spending review. Έχουμε διάφορες ε, τοποθετήσει και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την κριτική κατά του πράσινου προσανατολισμού. Όχι κατά της ιδέας ε, επί της αρχής, αλλά κατά της πρακτικής εφαρμογής της. Κατά πόσον λειτουργεί ή όχι αυτός ο οικολογικός πράσινος προσανατολισμός. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω. Γι' αυτό πιστεύω ότι η νομική μας βάση για την ε, κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Κάποιοι μου λένε ε, ότι οι εκπρόσωποι των γεωργών ότι εντάξει μπορεί να δεχτούμε κάποια περικοπή αν υπάρχει απλοποίηση της διαδικασίας σε ό,τι αφορά την ε, κατάθεση αιτήσεων, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της σωστής χρήσης ε, για την επιδίωξη των κοινών κανόνων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και, το περιβάλλον και την ε, γεωργία και την εκτροφή. Εμείς διαβάσαμε διάφορες αξιώσεις για την περικοπή που πρέπει να γίνει στην ΚΑΠ, για την ε, ε, περικοπή 13% για την επιστροφή αρμοδιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα θεωρώ σωστά. Μία ενιαία αγορά, μία εσωτερική αγορά είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί όταν υλοποιηθεί από κοινού και υπάρχουν κοινοί κανόνες. Ο κατακριματισμό και η επιστροφή αρμοδιοτήτων σε εθνικέ δομές θεωρώ ότι είναι λάθο δρόμο. Η κοινή γεωργική πολιτική ήταν η πρώτη άλλωστε υλοποιημένη κοινωτική πολιτική μετά την ε, Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και πιστεύω ότι αυτό παραμένει απαράλλαχτο. Είναι πιο σωστό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ε, τις περικοπές, αυτό που είναι σαφές είναι ότι θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 10% οι περικοπές αυτές, όχι παραπάνω για το 2020 δηλαδή και για το πρόγραμμα το 2021. Και έτσι λοιπόν το παλιό στο καινούργιο πουδοπού θα έχουμε περικοπές μόνο 5-10%. Θα πρέπει φυσικά να δούμε πού θα γίνουν αυτές οι περικοπές. Πού θα υλοποιηθούν. Εδώ θεωρώ ότι η εθνική συγχρηματοδότηση δεν αποτελεί πραγματικά το μέσο γιατί αυτό θα ήταν εις βάρος προφανώς των ε, αγροτών σε φτωχές σε περιοχές. Και θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα σήμερα με τη σειρά του περισσότερη, όχι λιγότερη γραφειοκρατία. Το θέμα των ορίων. Θα πρέπει να το απαντήσουμε και αυτό. Το θέμα της ε, βαθμίας μείωσης ε, των ενισχύσεων ανάλογα με την, ε, το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα το εξετάσουμε και αυτό. Και τον Απρίλιο με τον συνάδελφο Χάουγκαν θα αποφασίσουμε και θα σας υποβάλουμε λοιπόν τη σχετική μας πρόταση. Το ποσοστό σφάλματος. σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων. Στην και πολιτική το ποσοστό αυτό είναι σχετικά χαμηλό. Να Νομίζω λοιπόν ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να δείξουμε το θάρρος και να έχουμε την τόλμη να μην αυξήσουμε τους ελέγχους. Το single audit να αναθέσουμε αυτούς τους ελέγχους σε μία υπηρεσία Αυτό θα ήταν μεγάλη ανακούφιση, ξέρετε, για τους ε, αγρότε. Αλλά σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι το ποσοστό σφάλματος ε, με λιγότερου ελέγχου ενδεχομένω να αυξηθεί. Εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τους νερού αγρότε, την καινοτομία και τις άλλες εξελίξεις πέρα από την ε, γενική υποστήριξη να υπάρχουν ξεχωριστοί κορβανάδε. Να υπάρχει και ένας κορβανά ε, για περίπτωση έκτακτη ανάγκη, σε περίπτωση κρίση, σε περίπτωση ζημίας, σε ένα τμήμα της αγροτική παραγωγή, σε ένα τμήμα των χωρών ενδεχομένω. Άρα δεν θέλω επανάσταση, θέλω μετεξέλιξη για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την επόμενη γεωργική πολιτική. Ένα τελευταίο σημείο, επιτρέψτε μου. Αν θέλουμε να ταχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος, τι κάναμε την τελευταία φορά λάθος, τι πήγε λάθος. Η Επιτροπή Μπαρόσο τον Ιούνιο του 2011 πρότεινε την, ε, το πολιτές δημοσιονομικό της πλαίσιο για 7 χρόνια. Στη συνέχεια δεν έγινε τίποτε άλλο. Δεν σημειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ούτε στο δεύτερο ήμιση του 2011, ούτε στο 2012. Η συζήτηση ξαναξεκίνησε το 2013 μόλις. Μέσα Δεκεμβρίου λοιπόν του 2013 η εκτελεστική, ψηφίστηκαν οι εκτελεστικοί κανόνες, οι οποίοι και δημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στην επίσημη εφημερίδα. Μέχρι τότε ή τα επιμελητήρια, οι ενώσεις ε, αγροτών, μέχρι να ενημερωθούν όλοι αυτοί και μέχρι να εφαρμοστούν όλα αυτά και να υλοποιηθούν σε νομοθεσία στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες μέχρι να γίνουν οι αιτήσει, μέχρι να καταρτιστούν οι αγρότες. Είχαμε φτάσει ετσίως την άνοιξη του 2015. Γι' αυτό λοιπόν τα τρία πρώτα εξάμεινα του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου ήταν χαμένα. Χαμένα χρόνια. Όταν λοιπόν ε, ο, ο νερός γεωργός θέλει να οργανώσει την, τα εκτροφία του, θέλει να αγοράσει ένα μεγάλο μηχάνημα και έχει μόνο 20% παλαιού κεφαλαίου. Χρειάζονται 80% πίστοση από την τράπεζα, δάνειο. Η φρεγγιότητα του λοιπόν θα εξαρτηθεί από τη γιαγιά του, από την πεθερά του, που θα αγγιηθεί γι' αυτόν, είτε από ένα κοινό ε, αγροτικό πρόγραμμα αν δεν μπορεί να του πούν ότι τα επόμενα 7 χρόνια ε, θα πάρει ένα εκτάριο τόσα χρήματα και αυτό θα είναι ουσιαστικά ίδιο κεφάλαιο, τότε θα λάβει το δάνειο. Θα μπορέσει να αγοράσει τη μηχανή, το μηχάνημα που χρειάζεται. Άρα, όχι το Δεκέμβριο του 2020, δεν πρέπει να, να ψηφίσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο τον Δεκέμβριο του 2020. Θα, το Μάιο, λοιπόν, θα υποβάλουμε την πρόταση για το πακέτο και θα ακολουθήσουμε τα σύντομα, τα επόμενα βήματα. Πρόκειται για το έκτη έκδοση του πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου. Πρώτη του ήταν το Ζακ Τελόρ το 88. Αλλά μετά πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πριν από την υλοποίηση τον Ιανουάριο του 2021 θα έχουμε για πρώτη φορά εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές. Είτε λοιπόν εμείς οι δύο πριν από τις εκλογές, εσείς και εμείς, θα κάτσουμε να το κοιτάξουμε αυτό πριν τις εκλογές ή θα φτάσουμε Δεκέμβριο του 2020 πρωτού ψηφιστεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο. Όσο πιο νωρίς ορίσετε τους συζητητές που αναλάβουν το θέμα, αν ξεκινήσετε 3 Μαΐου τις εργασίες σας παράλληλα με το Συμβούλιο, τότε μπορεί να έχουμε και μια ευκαιρία και για τους γεωργούς μας και για την υπετρό μας να υπάρχει σαφήνεια νομική βεβαιότητα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και αυτό θα είναι για όλους τους φορείς μεγάλο πλεονέκτημα και στο ΚΑΠ και στον ορίζοντα και σε όλα τα προγράμματα όπου χρειάζεται μακροπρόθεσμα ασφάλεια επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Από δύο λεπτά στους συντονιστές. Ε, στο 1,5 λεπτό θα σηκώνω το σφυράκι για να ξέρετε ότι πλησιάζει ο χρόνο μας. Τρία λεπτά θα έχει ο συγητής και οι σκιώδεις συγητές επίσης. Για να, και να σπάσουμε τη γεωργία για να χρηματοδοτήσουμε άλλα προγράμματα. Και χαίρομαι που υπάρχει για να και να σπάσουμε τη γεωργία για να χρηματοδοτήσουμε άλλα προγράμματα. Και Χαίρομαι που υπάρχει. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε. Στις 21 Ιουλίου έβγαλα δίπλωμα οδήγηση για τρακτέρ. Τα δημητριακά κόστιζαν το σήμερα όσο ο κόστος ήταν κατά στοιχεία του 61, θα είχαν 37 της το χρόνο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα χρήματα που ξοδεύουμε για την γεωργική πολιτική, όταν κατανέμουμε και να μην ξεχνάμε ότι πάνω από 40 εκατομμύρια θέσεις εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται με την γεωργία. Έχουμε λοιπόν πολύ καλά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τα χρήματα που δαπανώνται στη γεωργία και χαίρομαι ιδιαίτερα που παρουσιάζει στατική έτσι, αντιμετώπιση στη γεωργική πολιτική και θα Γιατί 4 και τέταρτο πρέπει να φύγει ο Επίτροπος. Οπότε μέχρι 4 και πέντε θα δεχόμαστε ερωτήσει. Ο κύριος ε, Αντρίο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε ε, για αυτά που μας είπατε. Ε, μάλιστα, όταν αναλάβατε καθήκοντά σα, είχατε πει στην αρκτήρια ομιλία τη ότι θα πρέπει να φάει και καταπολέμηση τη τρομοκρατία και έρευνα το ίδιο. Ε, η επιστηστική όμως επάρκεια και επιστηστική ασφάλεια επίσης ε, είναι θεμελιώδη. Και το, τα τρόφιμα έχουν άμεση επίπτωση στην ε, δημόσια υγεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν δημόσιες πολιτικές που θα συνοδεύουν την. Χρειαζόμαστε μέσα, κονδύλια, αν δεν αλλάξει ο προπολογισμό, θα μπορούσαμε στη Γεωργία να κάνουμε κάποιε απαραίτητε μετατροπέ στο να λαμβάνουν υπόψη για τον οικολογικό προσανατολισμό και, το, και τη δημόσια υγεία. Αν όμω με τον προπολογισμό, θα είναι πολύ δύσκολα να τροποποιήσουμε την στρίπα του χρηματοδοτικού κενού που θα δημιουργηθεί από τον Brexit. Επίσης είπατε ότι οι αγρότες χρειάζονται ασφάλεια δικαίου για να... και μια προβλεψιμότητα για να σχεδία περίπου 29 χρόνια σε αυτήν την Επιτροπή πάρα πολλά χρόνια. Ε, στις 14 Φεβρουαρίου στην παρουσίαση που έγινε για το Πίτερ και επίσης ε, προσφέρει πολλά άλλα αγαθά που δεν έχω το χρόνο να τα αναλύσω. Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται ε, υπολογιστό και τον Επίτροπο Έτιγκερ για την παρουσία του. Όπως είπατε και στην ομιλία σας κύριε Επίτροπε, με το νέο οποία χρειάζονται και νέε προτεραιότητε. Συμφωνώ. Οι πολιτικέ και τα τρέχοντα προγράμματα φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί. σω θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια εξυγχρονισμού και να ε, εξετάσουμε προσεκτικά ε, μήπως κάποια ε, στοιχεία θα πρέπει να διαγραφούν. Και ενώ σχεδιάζουμε τις νέες μας πολιτικές, δεν θα πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα απολογισμό ε, και να κρατήσουμε το status κουβό και σε αυτό να χτίσουμε τις προτεραιότητες. Και αν είναι να προσθέσουμε σε αυτά που ήδη έχουμε, να δούμε μήπως μπορούμε κάποια στοιχεία να τα αναθεωρήσουμε και μερικά ακόμη και να τα καταργήσουμε. Ερωτώ λοιπόν, Πώ είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε και να έχουμε τι ίδιε προποθέσει ώστε πριν συμφωνήσουμε στο νέο ΠΔΠ να είμαστε βέβαιοι ότι η κοινή ορική πολιτική υλοποιεί του στόχου που έχουμε, δηλαδή για την καινοτομία, για την επιστημιστική ασφάλεια, για τη βιωσιμότητα. Πρώτα αυτόν τον απολογισμό θα πρέπει να κάνουμε, αν η ΚΑΠ ανταποκρίνεται στου στόχου μα. Έτσι θα, έχουμε, θα, δώσουμε και μία θεμητή εξήγηση προς τους φορολογουμένους μας που προβληματίζονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ε, Η κυρία Σένερα. Καλά το ίδιο είναι. Είτε πριν είτε μετά. Δεν έχει διαφορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν να πω ότι εμείς θεωρούμε ότι στο ισχύον πλαίσιο είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε περικοπή των γεωργικών δαπανών. Μια και τώρα όμως συζητούμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, κρίνουμε ότι το πιο σημαντικό, το Ποιο σκόπιμο θα ήταν πρώτα να προσδιορίσουμε τη νέα ΚΑΠ και μετά να δούμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες και να προσδιορίσουμε τον προϋπολογισμό που χρειάζεται για να εφαρμόσουμε την επιπλέον δημόσιες ενισχύσεις για τους γεωργούς, αν τα γεωργικά προϊόντα έχουν δίκαιες τιμές παραγωγού. Επίσης, μιλήσατε για την ανάγκη μείωσης, μια και αυξάνονται οι δαπάνες. Εγώ θα προτιμούσα αντί να μιλάμε για μείωση, να μιλάμε φορά που φεύγουν. Αν καταπολεμούσαμε τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, θα είχαμε αύξηση των φορολογικών εσόδων, οπότε δεν θα χρειαζόταν τόσες πολλές περικοπές. Και καλό θα ήταν ε, να μην αυξήσουμε, αλλά να μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες ή τις δαπάνες που στόχο έχουν... Περικοπές, αλλά είπατε ότι χρειαζόμαστε και πιο πολύ ε, αύξηση των εσόδων. Ε, εκεί θα πρέπει να στραφούμε. Αλλά είναι σαφές ότι θα μειωθούν τα κονδύλια. Αυτό δεν υπάρχουν αυτοπάτες δεν τρέφουμε αυτοπάτες Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι όταν μιλάμε για είναι πολύ πιο ουσιαστικό από το να μιλάμε μόνο για την πρώτο πυλώνα. Να υπάρχει μια ισορροπία δηλαδή, γιατί πολλοί ε, ανησυχούν ότι θα υπάρχουν υπερβολικές ε, περικοπές στο δεύτερο πυλώνα και ότι θα παραμείνει ο πρώτο πυλώνα όσο έχει ουσιαστικά. Ο πρώτο πυλώνα λοιπόν και οι πληρωμέ ε, στο πρώτο πυλώνα θα πρέπει τη βιοπικιλότητα να τονίσουμε το σκέλο του κοινού, της κοινή ωφέλεια, Να δώσουμε αυτή την εξήγηση δημόσια. Στόχφατημένη λοιπόν διάθεση των πόρων. Θα είχαμε δυνατότητα να κάνουμε και περικοπέ. Ε, μιλάτε για ανώτατα όρια, θα πρέπει εκτάσει και να μιλήσουμε και για σταδιακή μείωση. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω επίσης που μιλήσατε κατά της ε, επιστροφής στο εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ο φόβος μας ο μεγάλος. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή κοινή πολιτική. Και θα πρέπει λοιπόν να μείνουν στις Βρυξέλλες αυτά. Ο κ. Σαγνιώ. Ευχαριστώ. Συζητούμε το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και τι πρόσεξα. Στους ίδιους πόρους, εκεί το κομματάκι. Ίδιοι πόροι. Τα χρήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλήγει από του φορολογούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα κράτη-μέλη δεν έχουν κανέναν έλεγχο επί αυτών. Με μεγάλο ενδιαφέρον είδα πόσο τολμηρό είναι αυτό. Αυτή η πρόταση ε, ε, φόρο επί του άνθρακος επί των εταιριών, επί χρηματοδοτικών πιστώσεων φόρος, επί του ηλεκτρικού ρεύματος, επί καυσίμων οχημάτων φόρος, Οπότε ο καημένο αυτοκινητιστή παντιοτρόπω φορολογείται, έχει ΦΠΑ, κάτω μέλο τον φορολογεί, παίρνει από το ΦΠΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά νέα στα καύσιμα φόρο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και φόρο άνθρακα, που ίσω και αυτό να εφαρμοστεί. Πολύ τολμηρό, πάρα πολύ τολμηρό. Και για αυτού στη Βρετανία που θέλουν να συνεχίσουν να, μην, να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω θα πρέπει να το ξανασκεφτούν βλέποντα αυτό το πακετάκι. Εάν ήμουν στη θέση σας, και προσπαθούσα να μαζίσω αυτά τα χρήματα, γιατί να μην δείτε να πάρετε ένα κομμάτι από το ΦΠΑ. Το 1 τρίτο, το 1% παίρνετε από το ΦΠΑ που συλλέγεται. Αυτό είναι το προηγούμενο που υπάρχει. Γιατί δεν το ανεβάζετε στο 1% κάτι παρεμφερέ. Νομίζω ότι είσαστε τολμηρότατο. Και νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραν και θα σα χτυπήσει αυτό στι επόμενε εκλογέ. Οι υπουργοί εκεί, οι αρμόδιοι, επιμένουν και το 1,0% ενώ όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί και όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι υποδεικνύουν ότι δεν βγαίνει πλέον ε, το 1,0%. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή αυτή η στάση και αυτό το, παρ, το παρατηρώ όλο και πιο συχνά τις τελευταίες εβδομάδες ως στάση. Διαπιστώνουμε επίσης το εξή και αυτό το το παρατηρώ όλο και πιο συχνά τις τελευταίες εβδομάδες ως τάση. Διαπιστώνουμε επίσης το εξή. Η εδώ θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την νομική βεβαιότητα. Συμφωνούν και ένα από τους λόγους που φεύγουν είναι και αυτό. Αλλά εγώ είμαι υπέρ των ιδιών πόρων. Και μακάρι η Ισπανική κυβέρνηση ήταν πιο δραστήρια, πιο προαρατική δεν μπορεί να λέει κανείς ότι θέλει να παραμείνει χωρίς περικοπές ή κάπ και παρόλα αυτά να μην προβλέψει νέου ή να μην ταχθεί υπέρ νέων ιδιών πόρων. Επίσης έχουμε αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις. Μόλις ολοκληρώσαμε τον κανονισμό Omnibus και αυτό τροποποίησε την ΚΑΠ. Τώρα ε, σε λίγο θα χρειαστεί να κάνουμε και άλλη μεταρρύθμιση, περισσότερο λόγω δημοσιονομικών ε, κριτηρίων παρά τροποποίηση των στόχων. Χρειαζόμαστε ασφάλεια και από τις σημαντικότερες αλλαγές που χρειάζεται η ΚΑΠ είναι να μας ε, στοιχίσει το Brexit, το χρηματοδοτικό κενό. 30% περίπου από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχει η Γεωργία. Ε, και από αυτές τις περικοπές είπατε τελικά θα φτάσουμε σε 3,5 δισεκατομμύρια λιγότερα κονδύλια στη Γεωργία. Πώς όμως σκεφτήκατε το, το Brexit. Νομίζω ότι μπορείτε σήμερα να μας το εξηγήσετε και ίσως να δείξετε μεγαλύτερη γενοδορία σήμερα. Ο Βάιτσε, κύριε Επίτροπε, στην ε, παρέμβασή σα αναφέρετε κάποια θέματα. Το θέμα τη οικολογία, το μάλλον δεν αναφέρετε κάποια θέματα όπω η οικολογία, όπω η προστασία του κλίματο. Όπω ξέρετε, πρέπει να προστατεύσουμε την, ε, το κλίμα και μέσω την ανάπτυξη τη υπαίθρου και μέσω τη γεωργίας μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ούτε το θέμα τη υγεία το αναφέρετε. Η ποιότητα των τροφίμων έχει να κάνει προφανώ άμεσα με την γεωργία. Και επηρεάζει προφανώ ε, την υγεία του κόσμου. Το θέμα και επίση των θέσεων εργασία. Ο συνάδελφο από τη Μεγάλη Βρετανία το είπε ότι κάθε χρόνο χάνονται χιλιάδε δεκάδε. χιλιάδες θέσει εργασία στον τομέα του Άρα να τεθεί ο στόχο να διατηρηθούν οι θέσει απασχόληση και να δημιουργηθούν και νέε. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σήμα προ τι περιφερειε. Ένα τελευταίο θέμα, γιατί είμαι πράσινος ε, και θέσεις απασχόλησης και να δημιουργηθούν και νέες. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σήμα προς τις ε, περιφέρειες. Ένα τελευταίο θέμα, γιατί είμαι πράσινος ε, και... Για περικοπές μιλάει ο Επίτροπος και αυτό με τρομάζει. Εγώ θα μιλούσα για οικονομίες. Θα προσπαθούσα να αλλάξω κάπως την οπτική γωνία και την προσέγγιση. Περιθώρια για να γίνει αποτελεσματικότερη παρέμβαση και να υπάρξει εξοικονόμηση, εγώ θα εγκατέλειπα το δρόμο των περικοπών. Όπως ε, ήδη σημειώθηκε, 12 με 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κενό από το Brexit και νομίζω ότι... Ο κύριος Βαλκάρσελ, Σίσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας ε, σε αυτή την ανταλλαγή απόψε για ένα θέμα τόσο σημαντικό για τους αγρότες μας. Γνωρίζουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει αύξηση του ισχύτος προϋπολογισμού από το 1% στο 1,1 ή 1,15%. Αλλά γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνουν περικοπές στο γεωργικό προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, γιατί ε, οι δύο πολιτικές ε, είναι κύριες σημασία για να μειώσουμε τις ανισότητες, να ενισχύσουμε την ανάπτυξη πέθρου και να κρατήσουμε τον ε, πληθυσμό στις ε, αγροτικές ζώνες. Οπότε θα ήταν ολέθρια μια απόφαση περίκοπης του γεωργικού προϋπολογισμού. Ήδη οι γεωργοί πληρώνουν τα σπασμένα του ρωσικού εμπάργου. Δεν πρέπει να πληρώσουν και οι γεωργοί μας τα σπασμένα του Brexit, δεδομένων στις κρίσεις που αντιμετώπισαν για τις τιμές, τη γαλακτοκομική κρίση, την κρίση στο χείριο κρέας ή στα απορροκυπευτικά. Διαρωτόμαστε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται καθόλου να συγχρηματοδοτήσει τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ και όντως σκέφτεται να περικόψει κατά 15 έως 30% το γεωρικό προϋπολογισμό. Σοβαρά το σκέφτεται ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Φαίνεται ότι δείχνεται ποια είναι τα προβλήματα. Και είναι σημαντικό να δούμε πού θα λάβουν χώρα οι περικοπές. Διότι άμεσες πληρωμές δεν μπορούν να περικοπούν. Αντιθέτως, μάλιστα, Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να προσπαθήσει να εναρμονίσει τις άμεσες πληρωμές, διότι γνωρίζουμε ότι χώρες από την Ανατολική Ευρώπη έχουν χαμηλότερες πληρωμές αλεύσεων. Διαφορετικά δεν μπορούν να επιζήσουν χωρίς βοήθεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος κάτι εξίσου σημαντικό, να μην ότι... Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Θεωρώ ότι η ΚΑΠ είναι μια πληρωμή που κατατίθεται από την κοινωνία προς τους γεωργούς για να παράσχουν υπηρεσία σε όλους μας. Τουλάχιστον αυτό έπρεπε να είναι. Πληρώνουμε τους γεωργούς ότι στην Ευρώπη έχουμε τα πιο ποιοτικά τρόφιμα στον κόσμο, ότι παράγονται αυτά και είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές σε ανεκτές τιμές και διατίθενται με ασφαλή τρόπο, είναι ασφαλή τα τρόφιμα και έτσι εξασφαλίζουμε και την προστασία των γιών μας και των εκμεταλλεύσεών μας και εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει κάποια προσέγγιση σωστή για το κλίμα, για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του πέθρου. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η ΚΑΠ έγινε μια αποζημίωση, αντιστάθμιση, διότι οι γεωργοί δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής και γίνεται κάτι σαν επιδότηση προς τους και στους χονδρεμπόρους τελικά. Εάν πρόκειται περί υπηρεσίας, πρέπει να διερωτηθούμε. Περιμένουμε να έχουμε την ίδια υπηρεσία το 2020 με τα ίδια λιγότερα χρήματα από ό,τι πριν. Αυτό είναι ανέφικτο και απαράδεκτο εσείς τελικά υψώσατε ε, ε, μια ιδέα σαν αετό, είναι ευθύνη δική μας και των άλλων να τον ρίξουμε τον αετό σας. Αν θέλετε να κάνετε οικονομίες και θέλετε να κάνετε οικονομίες, κάντε το από αλλού. Έχετε μανία πανάτε δισεκατομμύρια για τον χρημάτων των φορολογουμένων για στρατιωτικά προγράμματα. Να τα περικόψετε από εκεί και όχι από τους γεωργούς. Αν κάθε μιλητής παραβαίνει κατά έστω και 20 δευτερόλεπτα το χρόνο αγόρευσης, δεν θα προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπατε και σωστά ότι η Επιτροπή μας ήταν κατά κάθε περικοπής της ΚΑΠ. Αληθεύει τουλάχιστον αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, η ΕΠΑ, η Κίνα και άλλοι, συνοδεύουν, δίνουν μεγαλύτερη υποστήριξη στις χώρες του στη Γεωργία. Και το δεύτερο, που συνεπάγεται από το πρώτο, το άνοιγμα των αγορών στην περίπτωση των διαπραγματευτικών των, των εμπορικών των διμερών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του Καναδά, ΗΠΑ, Μερκοσούρ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, αυτό το άνοιγμα είναι ει βάρο της γεωργίας συστηματικά και κυρίω τη κτηνοτροφίας μα. Και δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί. Όλα αυτά σορευμένα. Η ευρωπαϊκή γεωργία και ο κόσμο τη υπαίθρου κινδυνεύει να αντιμετωπίσει δυσκολίε με όλε τι συνέπειε οικονομικέ, κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ και υγεία που έχουν αυτά. Οι συνομοθέτε που είναι το Συμβούλιο, θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Επίτροπε, και εσεί θα πρέπει τελικά να το λάβετε αυτό υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριος Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για αυτά που μας είπε. Ε, αναφέρατε πολλά νούμερα, πολλούς αριθμούς και σίγουρα σε κάθε επιτροπή ε, ακούτε ότι τα μέλη θέλουν να διατηρήσουμε τον ισχύοντα προπολογισμό για να μην να τον αυξήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ενισχύσει στη Γεωργία, οι ενισχύσει αποτελούν ένα θεμελιώδη στοιχείο όχι στήριξη μια δραστηριότητα, αλλά στήριξη του γεωργικού εισοδήματο. Πόσε γεωργικέ εκμεταλλεύσεις δεν θα είχα βάλει λουκέτο χωρί τι ενισχύσει τη κοινή γεωργική πολιτική, Ε, μερικοί επικρίνουν την ΚΑΠ. Αλλά τα κονδύλια της ΚΑΠ εξασφαλίζουν το γεωρικό εισόδημα για πολλές οικογένειες και στην πατρίδα μου. Πολλές γεωρικές εκμεταλλεύσεις ε, λαμβάνουν περισσότερες ε, ενισχύσεις ε, από ότι έχουν εισόδημα για να εξασφαλίσουν το προστοζήν. Οπότε δεν έχουμε ίδιου είδους ενισχύσει στην ΚΑΠ με τις υπόλοιπες πολιτικές. Και μάλιστα μείωση κατά 7% του γεωρικού προϋπολογισμού θα οδηγήσει με βάση τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμών σε μείωση 8,2% του γεωργικού εισοδήματο. Ε, τα γεωργικά εισοδήματα είναι περίπου το 50% των εισοδημάτων των άλλων ε, επαγγελματιών. Πώς λοιπόν θα κρατήσουμε ε, ασφαλές και υψηλό το γεωργικό στα ίδια. Να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας, γιατί ε, επανειλημμένω έχουμε συναντηθεί και έχουμε μιλήσει, γιατί είμαι μέλο και τη Επιτροπή ε, Προπολογισμών και εκεί μα είπατε ότι το χρηματοδοτικό κενό του Brexit θα πρέπει να γεβηρωθεί από αυξημένε επιβροκοπέ. Ο κύριο Σεκέρσκι σα έκανε έναν υπολογισμό. Ακόμη και λάβουμε υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κενό του Brexit ε, είναι δεδομένο και θα καλυφθεί από την ΚΑΠ με 15-30% μείωση φτάνουμε σε 3,5 δισεκατομμύρια διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων στα τωρινά επίπεδα και στο επόμενο ΠΔΠ. Ενώ ε, είπαμε ότι θα γίνει μια εξομοίωση των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των παλιών και νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εσείς τι γνώμη έχετε για αυτήν την εξομοίωση. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις προσπάθειες που καταβάλατε να διαφυλάξετε την ΚΑΠ και την πολιτική συνοχής, κάτι που αναφέρατε. Σε προηγούμενη συνεδρίαση στο Στρασβουργό, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος είναι απόλυτα αληθές, διότι χωρίς αυτές τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χωρίς την ΚΑΠ και την συνοχή θα αντιμετωπίσουμε άλλα προβλήματα. Να σε πιστήσω η προσοχή στην πολιτική πρασινίσματος. Δεν πήρε παραπάνω ε, χρήματα, αλλά αντιμετωπίζεται αυξη... Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση όσον αφορά τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Θα πρέπει οι φορεί να καταβάλλονται εκεί που παράγεται το κέρδος. Ευχαριστώ κυρία Ριμπέρο, Κύριε Επίτροπε, μας ζητήσατε μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ναι, καλή ελαστικότητα, αλλά όχι ει βάρος τη γεωργία και όχι με περικοπές στο γεωργικό προπολογισμό. Σε αυτή τη φάση το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρουν εναλλακτικού τρόπους χρηματοδότησης του κοινοτικού προπολογισμού. Και με τι εναλλακτικέ αυτέ λύσει να αντιμετωπίσουμε και να αντισταθμίσουμε τα προβλήματά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση που στην καλύτερη περίπτωση διατηρεί το γεωρικό προϋπολογισμό στα τωρινά επίπεδα και στη χειρότερη τον μειώνει κατά 30%. Ενώ για το έρασμο. Plus ε, ή τον ορίζοντα 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης. Γιατί λοιπόν στη Γεωργία συγκεκριμένα προτείνεται τέτοιες περικοπές, μια και έχουμε όλο και νέες υποχρεώσεις και νέες απαιτήσεις από τους γεωργούς, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ ας σεβαστεί την σχεδόν ομόφωνη θέση της ε, Επιτροπής Γεωργίας που απέτησε για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον ε, διατήρηση της, ε, της, της του τωρινού επίπεδου του γεωργικού προπολογισμού. Ε, κυρία Χόιμπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που εκφραστήκατε έτσι για την κοινή γεωργική πολιτική. Έχετε δίκιο. Είναι η πρώτη πραγματικά κοινή πολιτική. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ οι εθνικοί προπολογισμοί σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή δηλαδή ευρωπαϊκούς, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει να τα έχουμε λοιπόν υπόψη μας αυτά. Και οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι έτοιμοι να συμβάλλουν τα απαραίτητα στον, εθνικό, στον ευρωπαϊκό κορβανά. Να έχουμε υπόψη ναι, επίσης για τους ε, νέους γεωργούς ότι δεν χρειάζεται μόνο μία υποστήριξη στην εκκίνηση αλλά και τα πρώτα χρόνια σε ό,τι αφορά την ανακατονομή. Εδώ θα πρέπει να εστιαστούμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μία κοινωνικά αποδεκτή γεωργική πολιτική σε ό,τι αφορά την εκτροφή για παράδειγμα χρειάζεται μεταρρύθμιση. Ξέρετε τι γίνεται στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίτρο Τρεις μου. Καταρχάς, πιστεύω ότι θα πρέπει να πολεμήσουμε για πιο πολλά έσοδα, πιο πολλά χρήματα. Θέλουμε δηλαδή, όπως αναφέρεται και στη Γερμανία, από πλευράς Γερμανίας έχει αναφερθεί ότι θέλουμε τέτοιους παραπάνω πορούς Κατά δεύτερον, οι γεωργοί θα αποδεκτούν τη διαδικασία την καινούργια αν αισθανθούν ότι είναι δίκαιη η μείωση. Αν η μείωση αφορά όλους. Η δεύτερη δυνατότητα, το 50-50%, το 80% και 20% αυτός ο τύπος. 3,2 δηλαδή δισεκατομμύρια περικοπές. Αυτό μπορούμε να το μεταδώσουμε ως μήνυμα στους γεωργούς. Και τρίτη παρατηρήση λέτε πόσα χρήματα έχουμε στην διάθεσή μας. Εμείς δώσουμε το hardware και το software θα είναι γεωργική πολιτική. Αυτή ήταν η συμφωνία. Σας υποστηρίζουμε λοιπόν. Ε, κύριε Επίτροπε, από τη μια μας μιλήσετε για το χρηματοδοτικό κενό του Brexit και από την άλλη για περικοπές, υπερβολικές περικοπές στο γεωρικό προϋπολογισμό όπως ε, επισήμανα και οι προλαλήσαντες. Μήπως το Brexit είναι το πρόσχημα για να περικοπεί ακόμη περισσότερο ο γεωρικός προϋπολογισμός γιατί όπως ε, είπαμε η κοινή γεωρική πολιτική είναι η πρώτη και σημαντικότερη ευρωπαϊκή πολιτική και η πρόταση για τον οικολογικό προσανατολισμό προκάλεσε θύελα κριτικών και επικρίσεων από τους γεωργούς. Φαίνεται ότι είναι παράλογος ο τρόπος εφαρμογής. Ε, επίσης, προτείνατε μία εξομοίωση των άμεσων ενισχύσεων στην Πολωνία. Οι άμεσες ενισχύσεις είναι πολύ χαμηλότερες από αντίστοιχες σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ε, και ενώ εδώ και καιρό μας υπόσχεστε τις, ε, την εξομοίωση των άμεσων ενισχύσεων, εξακολουθούμε στην Πολωνία να έχουμε χαμηλότερες άμεσες ενισχύσεις από τη γειτονική Γερμανία. Γιατί να έχουμε μερικέ χώρε υψηλότερε άμεσε ενισχύσει από άλλε. Θα πρέπει όλε οι χώρε να αναλαμβάνουν το ίδιο επίπεδο άμεσων ενισχύσεων. Κυρία Ρας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προασπίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική και πρέπει να παραμείνει ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική. Γι' αυτό έχουμε δύο κινδύνους να αντιμετωπίσουμε. Να περικόψουμε κονδύλια ή να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επικουρικότητα. Δεν θέλουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι' αυτό ζητήσαμε αύξηση των εθνικών συνεισφορών στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι μιλήσατε για το 1,1 μέχρι 9. Νομίζω ότι οτιδήποτε κάτω από το 1,3 το ακαθάριστο ε, χώρο προϊόντος των κρατών μελών θα ήταν ανεπαρκή συνεισφορά για να διαφυλάξουμε το γεωργικό προϋπολογισμό στα τωρινά επίπεδα. Θα ήθελα να είστε πιο φιλόδοξοι και να μιλάτε για 1,3 τουλάχιστον και πάνω γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια στον γεωργικό προπολογισμό. Επίση, για να αντιμετωπίσουμε τη, τη δημογραφική πρόκληση και τη γύραση του πληθυσμού ή την απερίμωση, θα πρέπει να διαφυλάξουμε την τωρινή γεωργική πολιτική. Μόνο έτσι θα κρατήσουμε νέου στην Ήπεθρο, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάγκη ίσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Νόιχλου. Σα ευχαριστώ. Τρει παρατηρήσει. Καταρχά, δεν υπάρχει πραγματική ε, κοινή γεωργική πολιτική. Έχουμε χώρες που έχουν κάνει σύνδεση από σύνδεση, έχουμε διαφορετική υπολογισμό αναέκταση. Αυτή η αξίωση ότι υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική με βρίσκει αντίθετη. Κατά δεύτερον, η αποτυχία της αγοράς. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί όπως κάνουμε τώρα και στο χειρίο κρέας και στο γάλα έχουμε μεγάλη αποτυχία. Αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε και να περιμένουμε τα, χρήματα της, ε, από τις Βρυξέλλες θα λύσουν τα προβλήματα, δεν θα τα καταφέρουμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς λειτουργεί πραγματικά η αγορά. Τρίτο, κύριε Ότιγκερ, θα σας θυμίσω ότι είπατε στην Ολομέλιο η μεγαλύτερη α, αδικία είναι στις γραμμικές α, ε, πληρωμές. Δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρχει αυτή η αδικία και θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους. Chair. Κύριε Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω τα στοιχεία σας και το έγγραφο ε, τροφοδοτούν μια πάρα πολύ ευρύ συζήτηση και αυτός είναι ο σκοπός. Δεν ξέρω γιατί 30% επελέγει ως πρόταση για περικοπές, αλλά άκουσα γεωργούς στην Ιρλανδία που θέλουν περισσότερα χρήματα από την ΚΑΠ για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα. Και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέστατο. Θέλω να ξέρω τα άλλα 22 κράτη-μέλη τι άποψη έχουν όσον αφορά τη θέση τους για την αύξηση των συνεισφορών στον προπολογισμό. Δεν θέλω να είμαι αρνητική, μεν. Μιλάμε για αυτό το θέμα σε σχέση με το Brexit. Όμω, απ' την άλλη, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι βολιδοσκοπήσει στον Ηνωμένο Βασίλειο όλο και περισσότερο τίνουν προ ένα σκληρό Brexit. Και αυτό θα επηρεάσει το γεωργικό τομέα πάρα πολύ σοβαρά. Και πράγματι, ίσω να πετύσει από εμά να δούμε αν πρέπει να αυξηθούν οι πόροι να εξασφαλίσουν τα μάλα, γι' αυτό το αναφέρω. Κύριε ε, Επίτροπε, από την κοινή γεωργική πολιτική υποφελούνται όχι μόνο οι αγρότες, αλλά όλοι μας. Γιατί ε, από τη στιγμή που η γεωργία παράγει τρόφιμα, οι καταναλωτές έχουν συμφέρον να είναι και να το εκτιμήσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα κονδύλια της ευρωπαϊκής πολιτικής που επαναλαμβάνω ε, ε ωφελεί όλους τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους γεωργούς. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, είμαι εδώ για να ακούσω τις απόψεις σας και να σχηματίσω εικόνα. Κοιτώντα τι λένε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Είμαι πραγματικά α, περίεργος κατά πόσον το, ήδη το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα πετύχει να συμφωνήσει. Το Brexit δεν είναι να έπε με μεγάλο αέχπε Αν φύγει λοιπόν αυτό το κράτος θα μας λείψουν 12-13 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθαρά. Αυτό είναι γεγονός. Και θα έχουμε και ένα λίγο ε, ασχολούμαι με γρίφους που μπορεί να λύσω. Άμα θέλετε εσείς να ανατρέψετε την πραγματικότητα, προσπαθήστε. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος. Πιστεύω ότι μια φιλόδοξη πρόταση θα πρέπει να υπάρξει, αλλά δεν θέλω στη συνέχεια να έρθουν τα κράτη-μέλη και να μας ε, τα πετακπάτε λοιπόν στο Άμστερνταμ και μιλήστε του. Τι επόμενε εβδομάδε στο Άμστερνταμ μπορείτε να πετύχετε πιο πολλά στο Άμστερνταμ για το σκοπό σα παρά εδώ στην αίθουση, πολύ περισσότερα. Καλή επιτυχία σα εύχομαι. Φυσικά δεν έχετε ε, τη μεγαλύτερη εγκύτητα με του συναδέλφου του ΕΛΚ, αλλά έχετε δικαίωμα να μιλήσετε. Καμία περικοπή στη γεωργία, καμία περικοπή στη συνοχή, πιο πολλά ε, μέσα για τη Σερβία, τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά θα πρέπει να ξέρετε σε τελική ανάλυση θα χρειαστούμε ομοφωνία. Θα χρειαστούμε 27 και παραπάνω εθνικά κοινοβούλια και αυτά θα χρειαστεί να συμφωνήσουν. Και έχω να σας πω ότι η διάθεση είναι δύσκολη. Θα το αποτύχουμε. Αλλά στην ομάδα σας μεταξύ μια ισχυρής ε, πολωνικής αντιπροσωπής και μιας μικρής γερμανικής υπάρχει ότι υπάρχουν αξιώσεις να μην υπάρξουν περικοπές για κάποια προγράμματα. Σε Erasmus Plus, για παράδειγμα, προτείνεται αύξηση αυτή. Η διπλησιασμός δεν θα είναι δυνατό, αλλά να υπάρξει αύξηση. Όχι. Αν η Ευρώπη θέλουμε να είναι ανταγωνιστική με την ε, Silicon Valley, με την Κίνα, θα πρέπει να δαπανίσουμε πιο πολλά στην έρευνα και την ε, καινοτομία. Θα πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας ε, πιο σωστά καταρτισμένες με το Erasmus Plus και τα παιδιά των ε, αγροτών θα πει να κάνουμε τα παιδιά μας ε, πιο σωστά καταρτισμένες με το Erasmus Plus και τα παιδιά των αγροτών θα ωφεληθούν από το Erasmus Plus αλλά υπάρχουν και ερευνητικά προγράμματα που είναι απαραίτητα για το γεωργό του αύριο ή το γεωργό του μέλλοντος. Γι' αυτό έχουμε και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Στη σωστή χρονική στιγμή. Και θέλω να πω ότι η κοινή γεωργική πολιτική φροντίζει για υψηλής ποιότητα στρόφιμα επαρκή εφοδιασμό και στην Ευρώπη και στην όλη την προστεθέμενη αξία των μεγάλων αυτών προγραμμάτων οι υπολογισμοί σας δεν είναι λανθασμένοι. Μιλάω για 5-10% μείωση και θεωρώ ότι είναι εφικτό αυτό. Αλλά ήδη στη δημοσιότητα έχουμε ακούσει πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής μια διαδικασία περισυλλογής, μια διαδικασία κατάρτισης ε, λευκής βίβλου θα είναι αξιόπιστη μόνο αν αναφέρονται όλες ε, οι απόψεις που ακούγονται στη δημοσιότητα. Εμείς δεν υφετούμε το 13% και το... Ο τύπος το 50-50% για την κάλυψη του καινού του Brexit την ε, παρουσιάζω σε κάθε ε, επιτροπή και σε κάθε ανακοίνωση τύπου και σε όλους τα ίδια λόγια λέω και στην κυρία Αρτού ε, χρημάτων. και αν θέλουν τα κράτη-μέλη να το καλύψουν, Α δώσουν 80% καινούργια χρήματα και 20% να γίνουν ανακατανομέ. Να γίνουν ανακατανομέ, μάλλον. Θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του κατά πόσο θα κάνουμε από εσά ε, να κάνετε προτάσει για περικοπέ. Αλλά σα παρακαλώ, αν ε, υπάρξουν ε, στοχευμένε περικοπέ, αυτό ζήτησε και ο πρόεδρο Γιούγκερ. Αν λοιπόν περάσουν τελικά ε, μα στον πραγματισμό προκειμένου να έχουμε την ελάχιστη ζημία και την μέγιστη ωφέλεια. Έφυγε ο συνάδελφος που μίλησε για τη σταδιακή μείωση των μεγάλων έργων. Ότι από την δική σας χώρα, τη Γερμανία και το ιστορικό της Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές φωνές που λένε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σημαντικός φορέας της οικονομίας και χρειάζεται υποστήριξη. Και ήταν ίδια στήριξη ανά εκτάριο, ίδιες άμεσες πληρωμές. Αυτό διακήρυξε. Ω εκ τούτου προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία θα πρέπει να έχουμε διάθεση να κάνουμε συμβιβασμούς, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει επιστηθέμενη αξία των τροφίμων για την ε, επισήμανση του τι περιλαμβάνεται μέσα στα τρόφιμα, στα κρασιά, στις συσκευασίε για την, την ε, Ιταλία, τυρί από την Γαλλία, όλα στην ίδια τιμή και με την ίδια ποιότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπιστούμε, να αγωνιστούμε. Όσο ποιες πολλέ κυβερνήσει μαζευτούν να καλύψουν το κοινό του Brexit Πλήρω. και όσο πιο πολύ λάβετε υποστήριξη ή κάποιοι αμήλικτοι που δεν θα θέλουν να δώσουν καθόλου παραπάνω χρήματα, θα παραμείνουν άτεκτοι στο 1,0% θα πρέπει να βρούμε διάμεσες λύσεις, 50%, 50%. Να ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο με ομοφωνία το επόμενο που τα επόμενα 7 έτη, θα προδώσουμε Όπως είπε ο κύριος ε, Επίτροπος, θα πρέπει να κάνουμε ε, διαβήμα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται τόσο σκληρές, σκληρές συνθήκες δεν καταφέρνουν να βγάζουν στο προς το ζήν. Η γεωρική πολιτική εξασφαλίζει... Ευχαριστώ. Είμαστε στο πλευρό σας πάντως. Ε, έχετε την συμπαράστασή μας. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστούμε και πάλι τον Επίτροπο. Ένα λεπτό γιατί μερικοί θέλουν να φύγουν από την αίθουσα. Ένα λεπτό διάλειμμα λοιπόν για να αποχωρήσουν όσοι θέλουν. E, e, Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Συγχωρήστε με γιατί ξέχασα να καλωσορίσω τους καλεσμένους του κυρίου Ρεμό από το Βέλγιο. Νέους αγρότες από το Βέλγιο. Ο Σεφ ε, χαιρόμαστε που παρακολουθήσατε ένα τμήμα της α, ε, συζήτησης που προηγήθηκε. Περάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Ο εισηγητής μας είναι στην αίθουσα. Ο δικός μας συντάκτης της γνωμοδότης είναι ο κύριος Νέκοφ. Κύριε Νέκοφ, επίσης ε, ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Πρώτα όμως ο κύριος Νέκοφ για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Η αγορά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι καινούριο και παρά τις πολλές πρωτοβουλίες που δρομολογήσαμε εμείς δεν είδαμε να γίνονται και αλλαγές στα προϊόντα που διατίθεται στους προμηθευτές. Σαν άνθρωπος που μεγάλωσε σε ένα από τα κράτη-μέλη που ενετάχθησαν προδεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας λέω με μιλότερη ποιότητα. Δεν αναφέρω μόνο στα τρόφιμα. Στα καλλιντικά, επίσης, σε διάφορα είδη μηχανημάτων στα αυτοκίνητα, στις υπηρεσίες. Σαν μέλος της Επιτροπής Γεωργίας πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε την κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων, στη δική μας περίπτωση. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα πρώτο βήμα και πιστεύω ότι θα έχουμε άριστο συντονισμό με τις άλλες επιτροπές, την Επιτροπή ΙΜΚΟ και την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Το σημαντικότερο πολιτικό μήνυμα είναι το ίδιο. Δεν είναι αποδεκτό στην ενιαία αγορά να έχουμε προϊόντα της ίδιας εταιρείας, της ίδιας μάρκας, με την ίδια συσκευασία, αλλά με διαφορετικά συστατικά, ποσοστά συστατικών, κάτι που είναι βλαβερό για χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κροατία κλπ. Σε κάποια κράτη-μέλη έκαναν έρευνες και είδαμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις όπου το ποσοστό κρέατος σε, σε κάποια προϊόντα είναι πολύ χαμηλότερο σε κάποιες χώρες από ό,τι άλλες. Στη Βουλγαρία επίσης είχαμε και άλλα παραδείγματα. Ένα προϊόν ήταν 107% πιο ακριβό στη Βουλγαρία από ό,τι το ίδιο προϊόν στη Γερμανία. Η τιμή ενός προϊόντος αποτελείται από πολλούς παράγοντες, διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Πολλοί από τους πολίτες μας προβληματίζονται διότι διαπιστώνουν ότι υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ μάρκας και ποιότητας. Αυτό που θα πρέπει να αλλάξουμε είναι αυτό με τη εμπορική πρακτική. Ένα προϊόν με την ίδια μάρκα να έχει την ίδια συσκευασία αλλά τα συστατικά να διαφέρουν. Συνάντησα κάποιους ε, προϊόν. και εκπλήσονται όταν βλέπουν διαφορά ποιότητας. Αν υπάρχει μια ντόπια συνταγή που είναι διαφορετική, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στην ετικέτα. Μια, ένα προϊόν από την ίδια εταιρεία με την ίδια συσκευασία έχει τα ίδια συστατικά ή τα ίδια ποσοστά συστατικών σε όλες τις χώρες. Αναφέρομαι, είναι το ταχύτερο δυνατόν αυτές οι έρευνες μέχρι το τέλος του 2018 και μετά να τροποποιηθεί η οδηγία που ανέφερα. Έχω και άλλες προτάσεις που πικά διάφορες τροπολογίες και θα ενδιαφερόμουν πάρα πολύ να γνωρίζω ποιες είναι οι απόψεις σας, ώστε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή θέση της Επιτροπής ε, Γεωργίας. Ευχαριστώ. Uh, Μάλιστα. 1,5 λεπτό οι και λεπτό. Ο κύριος Μπούντα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς ε, η πραγματικότητα είναι λυπηρή για μας για μας δηλαδή τους ε, πολίτες των ε, χωρών στις οποίες πολλούνται προϊόντα των ίδιων εμπορικών σημάτων αλλά με χειρότερη ποιότητα από ό,τι τα αντίστοιχα στις ε, υπόλοιπες χώρες. Είναι απαράδεκτο. Οι ίδιες μάρκες στη Γερμανία, η Ιταλία να έχουν καλύτερη ποιότητα από ό,τι στην Ανατολική Ευρώπη. Εντοπίστηκαν τέτοια προϊόντα μάλιστα από τις αρμόδιες αρχές και είπα ε, τοπικές συνταγές που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα τοπικά γούστα. Εδώ μιλάμε για τα προϊόντα του ίδιου εμπορικού σήματος που έχουν διαφορετική ποιότητα ανάλογα με τη χώρα στην οποία ε, πολλούνται. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούγκερ στην ομιλία του στο Ινολομέλεια για... Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω τέτοιου είδους φαινόμενα και να εφοδιαστεί με τα κατάλληλα μέσα για να θέσει ένα τέρμα σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές. Δεν μπορεί η ίδια εταιρεία να διαθέτει ε, προϊόντα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Νέκοφ για το σχέδιο γνωμοδότη. Σίγουρα οι πελάτες θα πρέπει, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, να ξέρουν τι αγοράζουν ε, στο σούπερ μάρκετ ε, σε όποια χώρα μέλος και αν βρίσκονται. Και φαντάζομαι η πλειοψηφία της Επιτροπής μας προτιμά να συστήνει στους καταναλωτές να αγοράζουν ντόπια προϊόντα για να να έχουν κάποια σχέση και με, το, με τη χώρα τους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, οι πολίτες ταξιδεύουν, οπότε όταν ε, ταξιδεύουν και βλέπουν το προϊόν από το ίδιο εμπορικό σήμα, περιμένουν να έχει την ίδια ποιότητα όπου και το αγοράζουν. Αν όχι 100% το ίδιο, θα πρέπει τα, τα συστατικά να είναι τα ίδια. Για να είναι σίγουροι ότι όπου και να αγοράζουν το προϊόν, από τη στιγμή που είναι του, του ίδιου εμπορικού σήματος, να έχει την ίδια ποιότητα. Μάλιστα το πρόβλημα έχει εντοπιστεί ιδιαίτερο στις ε, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Εκεί τα ίδια προϊόντα φαίνεται να έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή περισσότερα, ε, περισσότερα πρόσθετα. Το είδαμε επίσης και στην περιεκτικότητα κρέατος ε, κάποιων προϊόντων κρέατος. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή και θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ενημερώνεται καλύτερα ο καταναλωτής για τη σύνθεση των προϊόντων και επίση ε, να είναι βέβαιοι οι καταναλωτέ ότι εφόσον αγοράζουν το προϊόν έχει... Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω, να χαιρετήσω την γνωμοδότηση και να ευχαριστήσω τον ε, συντάκτη της. Το θέμα μας ενδιαφέρει άμεσα και υπάρχει και μια σάφια ταυτόχρονα. Δυστυχώς έχουμε την αίσθηση ότι είναι πολύ δύσκολο. Οι έχουν την τάση να παράγουν προϊόντα χειρότερη ποιότητα για την τόπια παραγωγή και να εξάγουν καλύτερη ποιότητα προϊόντα. Ο κύριο Ρέμπεγκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μια ένωση των ίσων. Δεν μπορούν αυτά να αποτελούν απλώς λόγια. Οι χρήστες, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν στοιχεία στη διάθεσή τους. Αυτά τα διπλά πρότυπα είναι ένα φορά σοβαρό ε, φαινόμενο, διότι είναι ένας μηχανισμός εξαπάτησης. Χρησιμοποιείται λοιπόν μια ετικέτα ψευδής. Υπάρχουν ήδη ε, μελέτες, υπάρχουν ήδη μελέτες που έχουν συνταχθεί από αυτού. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξουν δημόσιες πλατφόρμες στις οποίες οι ειδικοί και οι καταναλωτές των κρατών μελών να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τις ετικέτες και να κατορθώνουν να αντιπαραβάλλουν τις πληροφορίες που δίδονται στα προϊόντα που πολλούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. Έτσι είναι δυνατόν να ε, χτυπάει ένα συναγερμό αν υπάρχει πρόβλημα και να παρεμβαίνουν οι αρχέ. Και ο τρόπο θα είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστούν τα προϊόντα που είναι προβληματικά και οι πολίτε θα μπορούσαν έτσι να συμμετέχουν ενεργά στην λύση του προβλήματο. Ε, Το ο τρόπο θα ήταν δυνατόν ίσω να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία, ένα νέο φορέα, νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία και εκεί ε, βέβαια δεν θα υπάρχουν οι πόροι Όμω θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα των διπλών προτύπων. Ε, θα έλεγα ότι έχει συνέπειες στις κοινοτικές πολιτικές. Πώς να μιλάμε για νέα αγορά, όταν, πώς να μιλάμε για κοινέ αγορές και πολιτικές όταν έχουμε τέτοιες ε, περιπτώσεις σε επίπεδο 27 χρονών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 ε, ώστε να έχει επιρροή αυτή η έκθεση. Θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση όπως είπανε και οι προλαλήσαντες. Είναι κάτι παραπλανά και τους καταναλωτές ε, και που βλάπτει τους παραγωγούς. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτή η έκθεση και θα πρέπει να απευθύνουμε μια έκκληση της Γεωργίας. Ευχαριστώ κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον συντάκτη για την γνωμοδότησή του, γιατί πραγματικά επισημαίνει ένα πραγματικό πρόβλημα. Αλλά προσοχή, κάνουμε μια διάκριση. Έχουμε τα βασικά προϊόντα που διατίθενται με βάση συγκεκριμένες συνταγές με την ίδια συσκευασία. Και όταν εκεί είναι διαφορετική η ποιότητα, πραγματικά είναι σκανδαλώδες. Αλλά Πολλές φορές ε, και στην ίδια τη χώρα υπάρχουν διαφορετικά γούστα και ένας ε, παρασκευαστής ή ένας ε, διανομέας προσπαθεί να προσαρμόσει το προϊόν στο, στα γούστα της πελατείας. Πριν γίνω ευρωβουλευτής, ασχολήθηκα με την τυροκομεία και ξέρω ότι το ίδιο τυρί έχει διαφορετική γεύση ανάλογα με το σε ποια περιφέρεια διατί, διατίθεται. Αποκρίνεται το τελικό προϊόν στο γούστο του πελάτη που διαφέρει από περιφέρεια, από περιοχή σε περιοχή. Και σίγουρα τις τις πρακτικές θα πρέπει να τις εντοπίσουμε και να τις στυλιτεύσουμε και περιμένω σχετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αλλά σε ό,τι αφορά την προσαρμογή της αγοράς δεν θα πρέπει να τους βάζουμε όλους ε, στο ίδιο... Μόνο όταν το ε, πουλάνε στην Μεγάλη Βρετανία είναι στην δεξιά πλευρά αλλά είναι το ίδιο μοντέλο Audi. Αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ απλουστευτικό, αλλά αυτό για το οποίο παραπονιέστε είναι μια άλλη πτυχή του ίδιου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι κερδίζουμε, τι όφελο υπάρχει. Υπάρχει κάποια προβλήματα, του βάζουν χειρότερα υλικά και του χρεώνουν το ίδιο όπω θα του χρεώναν άλλο. Είμαστε δηλαδή απαταιώνε, αυτό συμβαίνει. Γιατί δεν άκουσα κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά τι τιμέ. Σε μια εποχή επιχειρηματιών. Υπάρχει δηλαδή μια παράλληλη μαύρη αγορά όπου πάει κάποιος δηλαδή στην... Λέει ο κ. ήταν παλιά μια χώρα. Αυτό συμβαίνει. Κάποιος βγάζει χρήματα σε μαύρη αγορά. Αν ε, δώσουν παραπάνω. Είπαν όμω κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Θα καλωσορίσω τον εισηγητή εδώ να είναι πολύ συνεκτικός και να δείξει πραγματικά επιμονή. Δεν είναι καινούργια αυτή η συζήτηση, ξέρετε, έγινε και ένας ε, συζητήσεων με τους ε, παραγωγούς, αλλά δεν είχαν ε, αποτέλεσμα. Αν θέλουν, μπορούν να το πετύχουν σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, ε, έχουν κάποιο ποτό χωρίς ζάχαρη, το βάζουν με μεγάλα γράμματα. Εδώ τι μας είπαν πολλοί οι πουλά ότι άμα θέλετε μπορείτε να διαβάσετε όλα αυτά αλλά αν ε, αγοράσω ένα προϊόν στην αγορά θεωρώ ότι αγοράζω την ίδια ποιότητα όπως όλο τον κόσμο. Αν όμως υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν διαφορές ανά περιοχή να το γράψουν. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που διαπιστώνω αλλά πραγματικά έχω εκνευριστεί γιατί αυτή η συζήτηση κρατάει χρόνια και δεν υπήρξε οποιαδήποτε νέα δέσμευση από πλευρά των παραγωγών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι καλό και πρέπει πραγματικά να δείξει επιμονή και να είσαι δυναμικός και σε ό,τι αφορά τους αυτοκινητο τη ε, της Γερμανίας δεν θα το διανοούντουσαν να δώσουν άλλη ποιότητα στην Αγγλία από ό,τι στη Γερμανία. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Εδώ κάτι με ανησυχεί και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάμε τα και να το κυνηγήσουμε. Γιατί το θέμα είναι τελικά να ενημερώνεται ο καταναλωτής αν το προϊόν χύψει. Ε, βάζει σιρόπι και όχι ζάχαρη. Έμα ε, να το χράψουμε. Αυτό προφανώς ε, δημιουργεί και ανησυχία και αντισπιστία στον καταναλωτή θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και να συνεχίσουμε να το κυνηγήσουμε το θέμα ε, και να είμαστε πραγματικά σκληροί. Θα πρέπει να τους κυνηγήσουμε τους ε, παραγωγούς. Σίγουρα. Ο καταναλωτής χαίρεται όταν ένα προϊόν ανταποκρίνεται στο γούστο του. Και από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αρκεί να υπάρχει σωστή επισήμαση και να ξέρει ότι κάτι απλώς ε, των προϊόντων, να κάνουμε κάποιες συστάσεις ε, στα κράτη-μέλη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε ε, τα προϊόντα του ίδιου εμπορικού σήματος να έχουν πατερικό ελέγχο. Αλλά και στα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε να πραγματοποιούμε ετησίως κάποιους εργαστηριακούς ελέγχους και ενδεχομένως των εργαστηριακών δεδομένων και να να δημιουργεί κοινέ βάσει δεδομένων. Θα δώσω τώρα το λόγο στην αρμόδια κατουσία επιτροπή για το θέμα αυτό, την Επιτροπή ΕΜΒ Η κυρία Όλγα Σέχναλόβα είναι η συντάκτρια του πονήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Μπίλιανα Μπόρζαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά μιλούμε για την ισότητα και τα ίδια δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα όπου δεν ισχύει ισότητα και τα ίσα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Που τη γνώμη έχουν όταν ε, έχουμε κατάφορες αποδείξεις ότι δεν ισχύει η ισότητα των πολιτών στην περίπτωση αυτή. Πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή θα δώσουμε και την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί του Ευρωπαίου πολίτε και στην πατρίδα μου την Κροατία 80% πρέπει να αντλήσουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έχουν γίνει πολλέ μελέτε για το θέμα αυτό και μάλιστα εγώ στην Κροατία, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων, με τον Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων, διαπιστώσαμε ότι και τρόφιμα αλλά και άλλα προϊόντα έχουν διαφορετική ποιότητα ανάλογα με την προτίμηση του παραγωγού παραγωγού να προσαρμοστεί στα γούστα του καταναλωτή και γι' αυτό το προϊόν μερικές φορές ε, έχει περισσότερα καρικεύματα, είναι πιο αλμυρό, λιγότερο αλμυρό, πιο ε, γλυκό, λιγότερο γλυκό. Ή τα αυτοκίνητα στην Βρετανική αγορά έχουν ε, το τιμόνι στα δεξιά, αλλά τα έχουμε κατάφορο παράδειγμα διακριτικής μεταχείρισης. Σκοπός μας λοιπόν είναι να συντάξουμε μια φιλόδοξη έκθεση ώστε να, να, βάλουμε τέτοιες πρακτικές στο μαύρο κατάλογο, στη μαύρη λίστα στην οδηγαστή συνεργασία και θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε έκθεση που θα μας καθιστά υπερήφανος. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ακούσαμε την κυρία Μπόρζαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Σέχναλοβα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ Προστασία του Καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Νέκοφ για το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς του. Μου άρεσαν οι παρεμβάσεις που άκουσα. Έχω ένα θετικό συνέστημα που δημιουργήθηκε τη συζήτηση. Έχουμε συντονιστεί, πιστεύω. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ ολοκληρώνει την έκθεση. Εγώ είμαι η και θα την παρουσιάσω τον Μάρτιο την έκθεσή μου. Οπότε περιμένω και τις δικές σας απόψεις. Και να υπενθυμίσω ότι το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα. Είμαστε στο 2018 και έχουμε έτοιμη την πρώτη κοινοβουλευτική έκθεση. Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Και έτσι θα συμβάλλουμε στην εξέβρεση λύσης. Διότι περιμένει πολύ καιρό να βρει λύση το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ε, εκπροσώπους από την Τζιγκρό και την Τζιγκάς. Δεν ξέρω, συνεννοηθείτε μεταξύ σας ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ. Και οι πρακτικές ε, που τονίζουν την τάση αυτή θα πρέπει γοργά να αντιμετωπιστούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ αρχής, όπως είπε, η Επιτροπή τι έκανε από τότε που ξεκίνησε για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτέ και για την ε, άδικη τις αθέμητες εμπορικέ πρακτικές ε, σε ό,τι αφορά την επί ελέγχου και δοκιμών για τα τρόφιμα που έχουν παρόμοια επισήμανση και παρούσα. Στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Σνέκοφ, υπάρχει και ένα πλαιτικό πρόγραμμα του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη ακριβώς της μεθοδολογία αυτής και το πρόγραμμα συνεχιστεί. Θα χρησιμοποιηθεί για να εξεταστούν και τα παράνομα αυτά προϊόντα. Και θα κοιτάξουμε και το σχέδιο έκθεση της κυρίας το Μάρτιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Να προσθέσω στα είδη υποθέντα το τον συνάδελφο του DigiGrow. Και εμείς προσπαθούμε Θέλουμε να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράσης στο λεπτομερές που δημιουργήσαμε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να τις ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα που έχουν για τους ελέγχους. Θέλουμε να τους στηρίξουμε. Ετήσεις για χορηγίες θα αξιολογηθούν μέχρι το τέλος Απριλίου για την υποστήριξη των αρμοδίων αρχών των κρατών Και όσον αφορά το, τη νέα συμφωνία, και σε εσά κύριε Πρόεδρε και στα συγκεκριμένα μέλη του Κοινοβουλίου ότι εξετάζουμε το θέμα αυτό που συζητείτε σαν τμήμα των σχεδιαζομένων τροπολογιών ε, των διαφόρων οδηγιών για, την, ε, για τους καταναλωτές, προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Ε, διαβλέπω πολύ καλής κατουσίαν επιτροπές ε, θα εκπονήσουν αξιόλογες εκθέσεις. Ε, ζητήσαμε ήδη αλλαγή νομοθεσία και θα πρέπει αυτό να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό και ε, είναι εύστοχο αυτό που μα είπε ο κύριο Νταντά ότι τα διάφορα τυριά έχουν και διαφορετική γεύση αλλά εκεί θα πρέπει να τη χάνουν προστασίες χάρη στην επισήμανση με την γεωγραφική προέλευση. Αλλά είναι άδικο να έχουμε στο ίδιο πακέτο το ίδιο προϊόν με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετικά υλικά. Ο κύριος Άγνιου έκανε μία ερώτηση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι γίνεται μια παραπλάνηση του καταναλωτή γιατί αγοράζει το προϊόν στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μια ιδέα για την ποιότητά του, μετά πηγαίνει στη Βουλγαρία, αγοράζει το ίδιο προϊόν και περιμένει να είναι εφάμιλο Αντίστοιχη ποιότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ετικέτας ή σήμανσης. Οι ετικέτες πρέπει να αντανακλούν ετικέτα η σήμανση οι ετικετες πρεπει είναι διαφορετική, η περιεκτικότητα είναι διαφορετική η περιεκτικότητα σε κρέας είναι χαμηλότερη στην Ανατολική Ευρώπη ή χρησιμοποιούνται περισσότερο. Αυτό όμω μπορεί να αποδειχθεί καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κάπω θα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε και έχουμε καραμέλα την έννοια τη αλληλεγγύη. Ε, θέλουμε λοιπόν αλληλεγγύη, ζώο ή το αντίστοιχο κινέζικο ανταλλακτικό. Ε, και τότε εγώ αποφασίζω, ο καταναλωτή, αν θα πληρώσω κάτι παραπάνω και θα βάλω το γνήσιο ανταλλακτικό ή θα προτείνω το επόμενο σημείο παρουσίαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Διεύθυνση, δηλαδή Άγκρη, για δείξει τη συντομογραφία, την επισήμαση και την παρουσίαση και σχετικά με την κατάρριση του κανονισμού τη Επιτροπή υπαριθμών 607 του 2009 ο κύριος Ζνούν για τις κατεξοδότηση πράξεις ε, στην ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς για να ετοιμάσει ε, με κατεξοδότηση πράξη με τρία κεφάλαια. Οι Υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνευσης με τα κράτη-μέλη, εκπροσώπους του αμπελονικού τομέα και άλλους ενδιαφερομένους στα πλαίσια της ομάδας πολιτικού διαλόγου. Και από τις σημαντικότερες παρακλήσεις που προέκυψαν από τις διαβολεύσεις ήταν η παράκληση, οι ετικέτες των κρασιών να πλουστευτούν, να γίνονται πιο ευανάγνωστες και να περιληφθούν σχετικές διατάξεις σε μια νέα νομοθετική πράξη. Ως εκ τούτου, η Γενική Διεύθυνση Άγκρη έχει ετοιμάσει μια ενιαία καταξιδότηση πράξη και την εφαρμοστική πράξη που καλύπτεται από τον κανονισμό 607-209. Η τελευταία ομάδα εμπειρογνωμόνων, στις 30 Ιανουαρίου, Εκεί και παρουσιάστηκε τελευταία εκδοχή του σχεδίου κατεξοδότηση πράξη που τροποποιήθηκε με βάση τα τελευταία σχόλια των κρατών μελών και τη γνωμοδότηση της νομική υπηρεσίας. Στη συνέχεια η ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, θα συνεδριάσει στις 17 Μαΐου, κατά την οποία και θα ψηφίσει ε, για την ε, εφαρμοστική αυτή πράξη, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη των κρατών μελών για το νομοθέτημα αυτό. Ε, μάλιστα, σε 7 Ιουνίου αναμένεται να εγκριθεί η ε, λόγω κατεξοδότηση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνέχεια θα μεταβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έγκρισή του από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Νοφρέ, που θα έχει 10 λεπτά το πολύ, για να μα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο κατεξοδότηση πράξη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με του βουλευτέ τη επίτροπή Γεωργία. Κύριο Νοφρέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κρυμμένοι ευρωβουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τελευταίο φάσμα προετοιμασία προτάσεω ευθυγραμμισμού του κανονισμού 607 για την κοιτοθεσία παρουσίαση, γεωγραφικέ ενδείξει και παραδοσιακού όρου στον τομέα του ίνου. Γίνονται διαβουλεύσει διάφορε υπηρεσίε και το κείμενο θα τηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επόμενου μήνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τα κράτη-μέλη. Και με εκπροσώπου των παραγωγών συνεργαστήκαμε κατανοούμε τις ανάγκες που υπάρχουν, τα συμφέροντα που υπάρχουν και πιστεύουμε ότι στο τέλος της διαδικασίας όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι ικανοποιημένα. Αποτελεί μας τη διαδικασία εφηγράμμισης της συνθήκη της αγώνας και της ε, δευτερογενού νομοθεσίας ε, του τομέα του ίνου που πρέπει να εξυγχρονιστεί. Είναι κρίσιμο αυτό για να αναπτυχθεί ο τομέας του ίνου και να έχει μια σωστή το να ανοίξουμε ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί ευκαιρίες. Μπορούμε σταδιακά να βελτιώσουμε τις διατάξεις με μικρορυθμίσεις. Στο σχέδιο κανονισμού συμπεριλάβαμε τις κάτωθι βελτιώσεις σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να χρησιμοποιούνται σύμβολα αποφεύγοντας τη χρήση γλωσσιμεγέθη των οσιών για αλλεργία, των διαφόρων γραμματοσυρών για αλλεργία και ο κανονισμό θα επιτρέψει μεγαλύτερη απλούστευση. Διαδικασίε για καταχώρηση και τροποποίηση των προδιαγραφών για τα προϊόντα έχουν ευθυγραμμιστεί με άλλου ε, τομεί των τροφίμων. Θα υπάρχει σαφή καταμερισμό να είναι το όριο για την εξέταση των αιτήσεων. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να εστιαστεί αποκλειστικά επί των βασικών στοιχείων του αιτήσεως σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεως και έτσι θα αποφύγουμε επικάλυψη εξέταση και ανάλυση. Ε, σε σχέση με αυτά που γίνονται ήδη σε επίπεδο κρατών μελών. Τέλο, οι παρού συμφωνίε όσον αφορά τα προϊόντα μα. Τέλο, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ αυτού του κανονισμού και τη ετικετοθεσία δια των τροφίμων και της αναφορά συστατικών. Μετά την έγκριση τη εκθέσεω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρτιο του 2017, ε, προσπαθήσαμε να ε, θέλαμε επεξεργαζόμενοι τον κανονισμό 607 να βάλουμε και άλλες πληροφορίες και συστατικά στην αντικειτοθεσία, να έχουμε ομοιόμορφη προσέγγιση και να μην έχουμε πολλαπλασιασμό των εθνικών μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί την προσέγγιση που είχε προταθεί, αλλά πιστεύουμε ότι οι δύο διαδικασίες είναι ξεχωριστές χωροχρονικά. Από τη μία πλευρά λοιπόν υπάρχει υποχρέωση η ετικοθεσία να αναφέρει συστατικά και διατροφικές ιδιότητες και απορρέει από τον κανονισμό για την προστασία των καταναλωτών και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τις γενικές διατάξεις για την ενημέρωση των καταναλωτών μέσω παρέκκλησης ε, της ε, δευτερογενούς νομοθεσίας, της παραγόγου νομοθεσίας. Επιλέξαμε από την άλλη ότι ο τομέας του ίνου χρειάζεται και αυτορύθμιση. Σε περίπτωση όμως που η αυτορυθμιστική προσέγγιση θα αποτύχει θα καθυστερήσει. Εν τη αυτή περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει διάφορες νομοθετικέ εναλλακτικέ λύσεις στα πλαίσια στα οποία μπορεί να κινηθεί. Τώρα μπορούμε να γραμμίσουμε